Bene, possiamo dare inizio alla nostra riunione. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Θέλετε το λόγο, τη συνάδελφε. Ha chiesto di parlare sul, sull'ordine del giorno. Έχετε κάποιο σχόλιο για την ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ. Δυνάμει το άρθρο 15 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι μετά από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβούλου παρουσιάζει την έκθεση των οποίων του Κοινοβουλίου. Όποτε γίνεται αυτό ε, στο διευρυμένο, στη διευρυμένη διάσκεψη των Προέδρων, ε, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί να μην την παρουσιάσει ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μόνο στη διευρυμένη διάσκεψη των Προέδρων. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε στο Στρασβούργο που διαθέτουμε και ημικύκλιο, γιατί ήταν πολύ αργά. Προτιμήσαμε λοιπόν ε, να, το κάνουμε αμέσως μετά το Συμβούλιο, κάνοντας χρήση αυτής εδώ της αίθουσας. Καταλαβαίνω Καταλαβαίνω, αλλά γνωρίζετε ότι το ημικύκλιο των Βρυξελών δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για όλο το χρόνο και για το 2013. Άρα έπρεπε να βρούμε μια διαθέσιμη αίθουσα εδώ στις Βρυξέλλες. Το σημαντικό είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάνει ένα απολογισμό των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα ήθελα εξ του Προέδρου Σούλτς να καλωσορίσω τον Πρόεδρο Φων Ρομπόη και τον πρόεδρο Μπαρόζο. Πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αυτό το οποίο ο πρόεδρος Σούλτς αλλά και μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών έχουν ήδη πει, δηλαδή ότι η πρόταση του Φόντρον Πόη για τη διαπραγμάτευση για μας είναι απαράδεκτη. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω μια επιθυμία. Ο πρόεδρος Φων Ρομπόη έχει ε, ένα τέτοιο ταλέντο διαμεσολαβητή, ώστε τις επόμενες εβδομάδες ελπίζουμε να μπορέσει να βρεθεί συμβιβαστική πρόταση που θα έρεται στο ύψος ε, των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, Ρομπέ, έχετε τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, Φυσικά θα έχετε ήδη λάβει γνώση των αποτελεσμάτων ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της, ε, προηγούμενη εβδομάδα. εβδομάδας. Δεν επετέχθη συμφωνία, μου ζητήθηκε όμως να προσπαθήσω να βρω συμβιβασμό, επειδή ε, φάνηκε ότι υπήρχε αρκετή πολιτική βούληση και σύγκληση θέσεων για να μπορέσουμε στις αρχές του επόμενου έτους να βρούμε μια συμφωνία, να καταλήξουμε σε συμφωνία. Βέβαια, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ουσιαστικά είναι θέμα για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται πάντοτε να το εξετάσει πληρώντας, εκπλώντας το ρόλο του δυνάμει του άρθρου 15 της συνθήκης. Δηλαδή, ε, καλείται να ορίσει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ένωσης. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει δυνατόν να επιτευχθεί συνένεση για το θέμα αυτό σε μία και μόνη συνεδρίαση, ούτε και στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν. Η ανάγκη ομοφωνίας βέβαια αποτελεί μείζωνα πρόκληση. Η εξέβρεση της συνένεσης απαιτεί ανταλλάγματα, δούνε και λαβίν και έναν κοινό, ε, μια κοινή αίσθηση σκοπού. Την εκτίμηση ότι από κοινού ορίζουμε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και δεν κάνουμε απλά μεμονωμένους ατομικούς υπολογισμούς για το πώς μπορούμε να ελιστοποιήσουμε τις εισφορές του κάθε κράτους μέλους και να μεγιστοποιήσουμε το τι λαμβάνει το κάθε κράτος μέλος. Ε, βεβαίως και αντιλαμβάνομαι τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες ε, του Κοινοβουλίου και έχω υπόψη μου και την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από τους ηγητές σας και από τις επιτροπές σας πολύ σωστά και πολύ επιδέξεις παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα τα σημεία τα οποία έχουν οριστεί από το Κοινοβούλιο ε, ε, συζητήθηκαν και πριν και κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι απόψει όμω του Κοινοβουλίου, όπω και οι απόψει τη Κομισιόν αλλά και καθενό ε, κράτου μέλου, θα πρέπει να εισαχθούν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ε, όπου η ανάγκη για ομοφωνία δημιουργεί κάποιους περιορισμούς ως προς την έκβαση. Ξέρετε ότι πρέπει να εργαστούμε πάνω σε έναν μετριοπαθή ε, προϋπολογισμό, γιατί αυτό απαιτούν οι καιροί. Είμαι, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέματα αυτά, διότι διατέλεσα υπουργό Οικονομικών και έχω αντιμετωπίσει τέτοια ε, προβλήματα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι είμαι ένας ε, απλός και ταπεινός απλά υπεύθυνος χάραξη πολιτικής. Απ' την άλλη πλευρά, σίγουρα στον προπολογισμό πρέπει να φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλουμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες μας, για τους πολίτες μας. Και η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να πράξει αυτά τα, ε, να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Και παρότι ε, Υπάρχουν περιορισμοί στους εθνικούς προπολογισμούς. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τομείς που μπορούμε δαπανώντα κάποια κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εξοικονομήσουμε χρήματα σε εθνικό επίπεδο, κάνοντα οικονομίε κλίμακα ή αποφεύγοντα επικαλύψει. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, που είναι κάτι το μοναδικό. Ξέρουμε ότι οι εθνικοί προπολογισμοί είναι συνήθως το 50% του ΑΕΠ, ενώ της Ένωσης μόνο το 1%. Σχετικά πολύ μικρός δηλαδή ο προπολογισμό. Ξέρουμε ότι είναι πολύ μικρός για την ε, διεξαγωγή μιας αντικυκλικής οικονομικής πολιτικής, αλλά σε κάποιες χώρες εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικός ε. κάποιε φορέ χρηματοδοτεί σχεδόν όλε τι δημόσιε επενδύσει και σε ορισμένου τομεί ε, επίση ε, σημαντικό όπω είναι έρευνα και ανάπτυξη και γεωργία. Άρα πιο πολύ αποσκοπεί στη διαρθρωτική οικονομική ανάπτυξη. Η κατάρτιση του παρόντο πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου ήταν διαφορετική από προηγούμενα αντίστοιχα εγχειρήματα και μια πιο δυσχερή διαδικασία. Πρώτη φορά όλα τα κράτη-μέλη συνειδητοποιούν ότι είναι η πρώτη φορά που δεν μπορούμε να περιμένουμε ανάπτυξη πραγματικού όρου. Επίση, για πρώτη φορά είχαμε 27 πλήρω συμμετέχοντε ε, με δικαίωμα νησικηρίας ε, που κάθισαν στο ίδιο τραπέζι. Φανταστείτε λοιπόν πω σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να καταρτιστεί προπολογισμό από τέτοιε συνθήκε. Επίσης, δεν ε, υπήρχε καμία προποφασισμένη συμφωνία μεταξύ μεγάλων χωρών. Και έχουμε και τον νέο ρόλο βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επίτευξη συμφωνίας είναι δύσκολη, όμω απαραίτητη. Θα απαιτηθεί πάντως περισσότερος χρόνος. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μια σύνθεση ε, σταθερότητας ε, και αλληλεγγύης. Πολλά θέλουν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να ενταχθεί στο πλαίσιο των γενικών προσπαθειών δημοσιονομικής συγκράτησης. Δεν συμφωνώ απόλυτα με την άποψη αυτή, διότι πιστεύω ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ουσιαστικά είναι ένας προϋπολογισμός επένδυσης. Βέβαια, αυτό αποτελεί και πολιτικό γεγονός που δεν πρέπει να ε, παραμελήσουμε και εγώ θα είμαι αυτός που θα πρέπει να βρω να αναζητήσω τη συμφωνία. Πρέπει να σας πω ότι οι δαπάνε όλα τα κράτη-μέλη πέστησαν μείωση κατά 1,5% του ΕΠ το 2011 μετά από θεαματική αύξηση που είχαν το 2008 και το 2009 Τη τάξη δηλαδή του 4 και 5 του ΑΕΠΑ. Όσοι λοιπόν ισχυρίζονται ότι οι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνονται στην πρότασή μου είναι εκτό θέματο, θα πρέπει να έχουν υπόψη τα εξή. Η πρόταση τη Κομισιόν τον Ιούνιο του 2011 ήδη περιλαμβάνει ονομαστικό πάγωμα στις δαπάνε για τη γεωργία και τη συνοχή, που συνολικά αντιστοιχούν στο 71% του συνόλου. 71%. Οι δικέ μου προτάσεις της 14ης και της 23ης Νοεμβρίου αντιπροσωπεύουν γενική συνολική μείωση 2% στους πραγματικούς όρου. Αν κανεί συγκρίνει μήλα με μήλα, δηλαδή μιλάμε για το σύνολο του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 με το σύνολο ε, του προγράμματος του 7-13. Παρ' όλα αυτά, στι προτάσει περιλαμβάνεται σημαντική αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη τη θέση εργασία και την ανταγωνιστικότητα σε σχέση με το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, που άλλωστε ήταν και η στρατηγική τη πρώτη Κομισιόν, την οποία και υποστηρίζουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε υπόψη μα την ανάγκη για περαιτέρω εξοικονομήσει πόρων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και το γεγονό ότι όλα τα άλλα τμήματα του προπολογισμού ανέρχονται στο μέγιστο ποσό των 280 δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν αποκλείεται ότι κάποιοι θα ήθελαν αύξηση των του 71 αυτού της 100. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση εγώ αρνούμε να αυτοσχεδιάσω. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρηθεί η αναπτυξιακή μας βοήθεια. Η πρόταση μου εξακολουθεί να περιλαμβάνει θετική ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Τώρα, στο επίπεδο των πόρων πρότεινα μεταρρύθμιση του ιδίου πόρου ΦΠΑ, να συμπεριληφθεί δηλαδή ο, ε, φόρος από τον χρηματοπιστωτικό συναλλαγό για τις χώρες που θέλουν τον εισαγάγουν, καθώς επίσης και προτείνω να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη στο σύστημα διορθώσεων. Το θέμα των πόρων είναι δύσκολο, είναι λεπτό και εμείς που πιέζουμε, μάλλον αυτοί που πιέζουν ε, για μεταρρυθμίσεις σε άλλους τομείς, δεν δείχνουν την ίδια διάθεση στον τομέα αυτό, τον ίδιο ζήλο και δεν έχουμε συμφωνία με όλους ε, τους καθαρούς ε, εισφορείς. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε και εδώ να βρούμε λύσεις, ίσως όμως λιγότερο φιλόδοξες. Η κατάρτιση του προπολογισμού πάντοτε υπήρξε πολύπλοκη διαδικασία και κατά το παρελθόν θα γνωρίζετε πολλοί από εσάς ότι δεν ήταν και το δημοσιονομικό πλαίσιο το 2015 μνημείο αισθητικής, δημοσιονομικής αισθητικής. Δεν θα πρέπει όμως να χαρακτηρίζουμε αυτή τη διαδικασία ως μάχη μεταξύ πλουσίων και φτωχών αγώνα μεταξύ βορρά και νότ. Η μισή περίπου από τις καθαρούς εισφορείς, μεταξύ αυτών και κάποιες μεγάλες χώρες, δεν έχουν ζητήσει διορθώσεις. Στο πλαίσιο της ομάδας αυτής, επίσης, δεν έχουν ζητήσει όλοι ακόμη περισσότερες ε, εξοικονομίες στον τομέα των δαπανών. Εδώ, μεταξύ των καθαρών αποδεκτών, σχεδόν κανείς δεν ε, ζητά αύξηση ε, των δαπανών όπως εγώ τις έχω παρουσιάσει. Επομένως νομίζω ότι η πρότασή μου μπορεί να στηριχθεί από πολλές χώρες, ακόμη και αν κάποιες από αυτές δεν είναι απολύτως ικανοποιημένε προς το παρόν. Αυτή η πολύπλοκη ε, ε, πραγματικότητα δεν μπορεί ε, με απλουστεύσεις να επιληθεί ή να συνοψιστεί. Θα επικεντρώσω λοιπόν τις προσπάθειές μου στην εξέβριση ενός δίκαιου συμβιβασμού δεν μπορούμε να μην ε, συμφωνήσουμε γιατί το κόστο θα είναι πολύ ψηλό για την Ένωση και για τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς εξαιρέσεις. Είμαι πεπισμένος, βασιζόμενος στο πνεύμα των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι αυτό είναι δυνατό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Βαν Ρομπόη και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μπαρόζο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Ευρωβουλευτές. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σας ενημέρωσε για τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πριν έξι μέρες είχα παρουσιάσει στο Στρασβούργο τη δικιά μας προοπτική, οπότε θα σας πω ποια είναι η αξιολόγησή μου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτού και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ κρατών μελών, ακόμη και αν πολύ. Ήθελα να συμφωνήσω στη συμβιβαστική πρόταση που παρουσίασε ε, η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμφωνία και θα πρέπει ακόμη να μπορέσουμε να καλύψουμε την καθυστέρηση που έχουμε, δηλαδή να καταρτήσουμε το MFF μέχρι το 2014. Δεν είναι όμως τόσο πολύ ο χρόνος που μας μένει. Και όπως είπα και την Παρασκευή το βράδυ, την περασμένη εβδομάδα είχαμε τις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις για το πολιωτές δημοσιονομικό πλαίσιο. παρόλο που η συζήτησεις αυτές έγιναν σε ένα πλαίσιο οικονομικής κρίσης και οι συζητήσεις ε, αντικατόπτριζαν αυτό το κλίμα. Παρόλα αυτά όμως έπρεπε ε, να ε, μπορέσει να υπάρξουν και επενδύσεις που είναι απαραίτητες σε περίοδο κρίσεως. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη θα υπάρχει ένα μικρότερο MFF διότι στο παρελθόν πάντοτε ε, υπήρχε συμφωνία και άμεση μετάβαση από το ένα ε, πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο στο επόμενο. Ενώ τώρα μιλάμε για περικοπές και είναι πολύ πιο δύσκολο να συμφωνήσουμε τις περικοπές από ό,τι, μπορεί από ό,τι είναι να συμφωνήσουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος αναπτύσσεται. Γι' αυτό και τώρα που η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις βλέπουμε ότι ορισμένες κυβερνήσεις ε, δεν ενθουσιάζονται με την ιδέα επενδύσεων προς ανάπτυξη. Λείπει λοιπόν η συνεκτικότητα. Πώς μπορούμε να είμαστε συνεπείς. Από τη μια μεριά λέμε ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις και ανάπτυξη και όταν φτάνει η κρίσιμη σημεία να πάρουμε τις αποφάσεις δεν ε, μπορούμε συλλογικά να προχωρήσουμε να απαντήσω σαφώς ότι η πρόταση που έχουν τώρα τα κράτη-μέλη στο τραπέζι ε, δεν συγκρίνεται με τα προηγούμενα δημοσιονομικά πλαίσια. Και όσον αφορά το θέμα της ε, δημοσιονομικής ολοκλήρωσης προσπαθήσαμε ε, να ε, καλύψουμε τις, τις πρόοδους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν στο πακέτο των έξι μέτρων που δεν διαμορφώνονται μόνο δραστηριότητες και αρμοδιότητες για τα θεσμικά όργανα ε, ε, αλλά ε, από κοινού για την Κομισιόν και τα θεσμικά όργανα. Και γενικώ τώρα υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μιλάμε για περικοπές. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις νέες αρμοδιότητές μας ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε νέες ευθύνες εάν μας ζητηθεί. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα θεσμικά όργανα όργανα της Ευρώπης δεν μπορούν συγχρόνως να αφαιρέσουν τα μέσα με τα οποία μπορούν να εκπληρώσουν αυτές τις ευθύνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε σε αυτή τη συνάντηση, διότι Ακόμη υπάρχουν σημαντικές διγνωμίες σε πολλά σημαντικά θέματα, ε, το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού και τη μορφή κατανομής μεταξύ των κρατών μελών. Συγχρόνως και πρέπει να είμαστε δίκαιοι προς τα κράτη-μέλη, κανείς δεν αμφισβήτησε ε, το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει ένα συμβιβασμός μεταξύ των 27, αλλά θα χρειαστεί περισσότερο καιρό μέχρι ότου να οριμάσουν οι αποφάσεις αυτές. Νομίζω ότι αυτό που διεφάνει σε αυτό το Συμβούλιο είναι ότι ο καθένας κατάλαβε καλύτερα τις θέσεις του ομολόγου του καθώς επίσης και τα συμφέροντά του και τα ενδιαφέροντά του. Ίσως όχι όλοι, αλλά νομίζω ήταν πολύ επικοδομητικό για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μία συνένεση στις επόμενες εβδομάδες. Κάποιος με ρώτησε πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε τις ε, θέσεις. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και για μένα είναι σαφές ότι όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε και οι καθαρά πληρωτές ε, και τα ταμεία συνοχής και άλλα και ε, το ταμείο για τη γεωργία και γεωργίας και ε, το μέσο για να συνδεθούν τα διάφορα μέρη της Ευρώπης και το Ταμείο Συνοχής και γενικά να υπάρχει συζήτηση, να υπάρξουν δύο ορθώσεις και ε, ε, όλοι συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών θεσμικών εργάνων θα πρέπει να κάνουν συμβιβασμόν. Η πρώτη δοκιμασία του εάν υπάρχει μία τέτοια συνένεση είναι ε, η δοκιμασία να δούμε αν θιοθετηθεί το προπολογισμό του 2014. Πλησιάζει το 2014 και δεν έχουμε προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν μπορεί να, υπάρξουν, να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο δημοσιονομικών ε, αρχών. Έχω μαζί με τον κύριο Βαν Ρομπόη συμμετάσχει σε συζητήσεις ε, σε όλες ε, τις, με όλες τις χώρες, 28 συμπεριλαμβανομένες και της Κροατίας. Ξέρω τι δέχεται και τι απορρίπτει ο καθένας, αλλά πιστεύω ότι θα πετύχουμε αν όλοι σκεφτούν πόσο ο καθένας μπορεί να προχωρήσει και τι είναι οι κινήσεις που χρειάζονται για να προχωρήσουμε. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει μία κρίσιμη μάζα για επενδύσεις και πρόοδο και επειδή η συμμετοχή στις δαπάνες επηρεάζει πολλά θέματα όπως η ελεύθερη διακίνηση ε, της ε, γνώσης, τον πολιτισμό, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική μας συνοχή θα μπορέσει να είναι ισόφιλος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ένα πνεύμα συνοχής για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ιδίως για τις πλέον απόμακρες περιοχές και χώρες της Ευρώπης. Θα είναι και ένας μοχλός για να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής η οποία πρέπει να προσφέρει και στην Ευρώπη και όχι μόνο στους γεωργούς τη δυνατότητα και του πρασινίσματος αλλά και τη διατροφική ασφάλεια για όλους. Επίσης ε, θέλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι με αυτούς οι οποίοι πλήττονται από την κρίση και να δεσμευτούμε ότι θα στηρίξουμε τους ασθενέστερους. Θέλουμε η πολιτική μας να είναι πιο δίκαιη και απλή Και αυτό προσπαθούμε να διατυπώσουμε. Να έχουμε επίσης μία αύξηση της αποτελεσματικότητας. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες οι οποίες ε, μπορούν να αποφευθούν Δεν εννοώ να μειώσουμε ε, το κόστος των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, διότι αυτό που δεν μου άρεσε ήταν η η συνεχής ε, επίπληξη ε, ε, και η κρίση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους διαδρόμους και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και λέω στους διαδρόμους γιατί στις συναντήσεις ήταν σοβαροί, ευγενείς, αξιοπρεπείς και πολλοί απάντησαν όταν τους έδωσα αριθμούς συγκεκριμένους για τα θεσμικά όργανα και ε, ε, επίσης ε, σεβαστήκαμε την, το fair play το οποίο πάντοτε ισχύει στις διαπραγματεύσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι μικρός. Το 2% από τον συνολικό προϋπολογισμό της Ενώσεως και πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και δύο ορισμένες κρίσιμες για όλα τα θεσμικά όργανα ε, έχω κάνει έκκληση για να υπάρξει ε, μία έγκυρη ε, δημόσια υπηρεσία στην Ευρώπη και επιμένω. Καταλήγοντας λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εξυγχρονίσουμε τον προϋπολογισμό μας, να εξηγούμε την συλλογιστική μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας εσωτερικά και προς τα έξω για την επόμενη εφταετία Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πρόοδο τις επόμενες εβδομάδες εγκαίρως για να υπάρξει μια συμφωνία έγκαιρη. Ευχαριστώ κύριε Μπαρόζο. Τώρα ξεκινάμε με τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων ξεκινώντας με τον κύριο Ζωζεφ Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, απογοητεύτηκα από τα αποτελέσματα της σκέψης κορυφής προηγούμενες εβδομάδες, διότι οι πιο σκεπτικιστές επέβαλαν τα άποψή τους στους άλλους ηγέτες και αντί να εργαστούμε προς το κοινό καλό, κάποιοι ηγέτες θέλουν να παίξουν το παιχνίδι της ε, ποιος είναι ο πιο δημοφιλής. Και θα επενδύσει τον James Clark. Η διαφορά μεταξύ ενός αργού κράτου και πολιτικού άνδρα είναι ότι ο πολιτικός άνδρας σκέφτεται τις, ε, ε τις επόμενες εκλογές και την εκλογή του, ενώ ο καλός πολιτικός άντρα και αρχηγός κράτους σκέφτε τι επόμενε γενιές. Ας σκεφτούμε τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η πρόκληση. Το... Αυτό το όραμα λείπει από κάποιους ηγέτε μας, οι οποίοι για να είναι αρεστοί στην κοινή γνώμη δεν έχουν το θάρρος να υπερασπιστούν την Ευρώπη για να βγούμε από την κρίση. Αλλά με κάποια ανακούφιση θα έλεγα και το εξή. Αν είχε ευρεθεί συμφωνία την ε, Παρασκευή θα ήταν κακιά συμφωνία. Καλύτερα λοιπόν να μην υπάρχει συμφωνία παρά να υπάρχει μια μέτρια συμφωνία. Η μείωση του προπολισμού σε 75% δι σε σχέση με την πρώτη επιτροπή είναι κάτι το οποίο σημαίνει πάγωμα του ευρωπαϊκού προπολισμού μέχρι το 2020 ε, σε ποσοστό 3 με 4 δις ετησίως και Καμία χώρα δεν έλαβε αυτή την απόφαση για τον εαυτό της, διότι πιστεύω ότι και τέτοιου τους προτάσεις δεν είναι υπεύθυνε. Η Ευρώπη δεν είναι μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών και αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτύχουν. Το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι μόνο προπολογισμό, είναι και μια πολιτική πράξη, η έκφραση μιας φιλοδοξίας παίρνουμε δεσμεύσει για να χρηματοδοτήσουμε κοινά έργα και πολιτικέ για ένα κοινό μέλλον. Χρειάζεται να το υπενθυμίσω. Όπω είπατε και εσεί, ο προγραμματισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 1% του συνολικού πλούτου τη Ευρώπη. Και αυτό το 1% χρησιμοποιείται σωστά. Και αν υπολογίσουμε τη συνεισφορά των συμπολιτών μα, όπω όλοι το έκαναν, και εμεί κάναμε του υπολογισμού μα, βλέπουμε ότι έχουμε αναμέρα και αναευρωπαίο πολίτη 64 σέντσα. Δηλαδή λιγότερο από ό,τι κοστίζει ένα καφέ εξπρέσο. Αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στα κράτη-μέλη υπό τη μορφή επενδύσεων στα έργα υποδομής, στην εκπαίδευση ή ως κονδύλια των διαθετικών ταμείων. Και αντίθετα από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο προπολογισμό, ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι 94% αποτελείται από επενδύσει. 4% μόνο αφορούν τι δαπάνε λειτουργίε και 2% ε, χρησιμοποιούνται για την μετάφραση και τη διερμηνία. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε κάθε μέρα. Οι 30.000 υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα τρίτων ε, των υπαλλήλων της εφορίας και των ε, ε, τελωνίων της αυτού μεγαλειότητας. Ειλικρινά λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τα κράτη-μέλη αφενός που επιβάλλουν όχι περισσότερες δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη κάνουν όλο και περισσότερο περικοπές στον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Στην ιατρική, ένας μόνο υπάρχει για τέτοιου είδους πρόβλημα Πρόκειται για διπολισμό. Διπολική προσωπικότητα λοιπόν. Το να προτείνουμε λοιπόν μείωση του προπολισμού για την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη σημαίνει ότι έχουμε πολύ κοτόφθαλμο όραμα. Όχι μόνο τα χρήματα τα οποία επενδύθηκαν θα απολεστούν, αλλά ακόμη πιο σοβαρό στέλνουμε πολύ κακό μήνυμα στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο όλοι λέμε ότι αυτό δεν είναι δική μας προτεραιότητα και σε δύο χρόνια ε, δραστηριότητας το ε, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας που άρχισε με startup και με πάρα πολλά ε, γραφεία ευρεσιτεχνίας δεν θα λειτουργεί σωστά, διότι κανένα σχέδιο, αν δεν είχαν δοθεί κονδύλια, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Το 2012 χρειάστηκαν πολλά ευρώ για να μπορέσουν να δοθούν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμους κονδύλια στα ε, ευρωπαϊκά κράτη. Ζητούνται 19 εκατομμύρια τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Χρειαζόμαστε αυτό το προπολογισμό και παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι πρέπει να υπάρξουν περικοπέ στον προπολογισμό. Πού υπάρχει η λογική. Θα σα δώσω και ένα τρίτο παράδειγμα. Θα πρέπει να επενδύσει περισσότερα από 1.003 σε έργα υποδομή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε αυτό το τμήμα για τα ηλεκτρικά δίκαια, για το ίντερνετ, για τα γραφεία, για το οδικό δίκτυο, για το σιδηροδρομικό δίκτυο που δεν πηγαίνει στην Μόσχα, αλλά προ τι Βρυξέλλε και τι άλλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσες. Και για κάποια κράτη-μέλη, στην περίοδο αυτή τη κρίσεως, πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία θα πρέπει να επενδυθούν. Γι' αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμεί με την ομάδα θα συνεχίσουμε να είμαστε υπέρ ενό πραγματοστικού και ρεαλιστικού προπολογισμού στο ύψο των προσδοκιών και των προκλήσεων. Πρέπει να πω ότι εμείς ενεργούμε συνεκτικά. Το πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή ε, είναι ελιστικό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα αγωνιστούμε όπως μπορούμε για να μην υπάρξουν περαιτέρω περιοχές. Πρέπει να σας πω ότι εμείς πρέπει να μπορέσουμε να αποφανθούμε με ενισχυμένη ψηφία. Η Ευρώπη βασίζεται στην ευημερία, στην ελευθερία, στην ελεγγύη. Πρόκειται για τρεις αξίες οι οποίες αποτελούν τη βάση των ιδανικών μας. Και έχουμε εδώ και την Επιτροπή, είναι θεματοφύλακα σε αυτόν τον αξιών. Πρόεδρε Βαν Ρομπόη, ποτέ δεν θα μπορέσουμε εμείς να αποδείξουμε αν δεν ενεργήσετε πάνω από τις αποφάσεις των κρατών μελών. Νομίζω ότι θα πρέπει για να υποστηρίξετε την ε, έρευνα και την απασχόληση να βρείτε τα κατάδια κονδύλιο. Χέρμαν, σου ζητώ να κάνεις ό,τι έκαναν πριν από 60 χρόνια οι πατέρες της Ευρώπης. Και πρέπει να σα πω ότι κανένα δεν θα σα εγκαταλείψει. Από κοινού θα αγωνιστούμε για να επιτύχουμε από κοινού. Και θα ήθελα να χαιρετήσω τη σοβαρή εργασία που επιτελείται από τον πρόεδρο Μπαρόζο και τι υπηρεσίε του που μα πρότεινε ένα ρεαλιστικό προπολογισμό και λαμβάνοντα υπόψη για την κρίση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητέ πρόεδρε Μπαρόζο, πρέπει και εσύ να αγωνιστεί. Πρέπει να περασπιστεί του ε, αξιωματούχου σου που εργάζονται. Θα ήθελα απλώ και μόνο να πω το εξή αρχίσουμε να κάνουμε συγκρίσεις. Ας δούμε τις, ε, πώς είναι η εθνική αξιωματούχη και πώς είναι η κοινοτική αξιωματούχη. Και με τη δουλειά που επιτελείται και με την αξία τους πάλι οι δικοί μας, οι ευρωπάλληλοι θα νικήσουν. Και πιστεύω ότι θα πρέπει το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο, αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να το παρατείνουμε το 2013 έως να ευρεθεί νέα συμφωνία για τους ιδίους πόρους που θα μας επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές που έχουν ήδη αποφασιστεί μειώνοντας και την εθνική συμμετοχή του καθενός. Και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών τα κράτη-μέλη θα σκεφτούν σοβαρά τις επιπτώσεις της κοντόφθαλμης αυτής πολιτικής που θέλουν να κάνουν. Και θα πρέπει να σκεφτούμε για τους πιο ευάλωτους από τους συμπολίτε μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τους στερήσουμε την, ε, τα ωφέλη του προγράμματος προς τους πιο ευαίσθητους και ευάλωτους. Νομίζω Ελπίζω ότι τον Ιανουάριο με τη νέα Προεδρή της Ιρλανδίας με... θα επικρατήσει το πνεύμα αλληλεγγύης και η επιστροφή στο ευρωπαϊκό πνεύμα για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ στον κύριο Ντόλ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Σβόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήταν ένα συμβούλιο στο οποίο δεν ελήφθησαν ε, αποφάσεις και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Αυτό όμως το οποίο δεν συμβιώνουμε και δεν δεχόμαστε είναι ότι πολλά μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να δεχθούν ότι και οι γυναίκες μπορούν ε, να υπάρξουν σε υψηλές ε, σχέσεις και θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την ισότητα των ανδρών με των γυναικών. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, τι ήταν ακριβώς αυτό το συμβούλιο. Ήταν ένα συμβούλιο όπου υπήρχαν εθνικισμοί και όπου υπερίσχυσαν οι εγωισμοί. Δεν ξέρω ποιος μίλησε για εν ονόματι ε, του ε, επικεφαλής ε, των κυβερνήσεων της Ευρώπης. Ο καθένας μιλούσε για τον εαυτό του. Και ήταν κάτι που δεν αξίζει στην Ευρώπη διότι πολλοί από εμά δεν αντιλαμβάνονται αντιλαμβάνονται ότι ε, μπορούν πρώτα να επηρεάσουν ε, την Ευρώπη περισσότερο αυτοί που έχουν αποστασιοποιηθεί και ότι ο Κάμερον ο οποίος σε δύο-τρία χρόνια μπορεί να μας πει αφήστε με να βγω από την Ευρώπη επηρεάζει περισσότερο την Ευρώπη σήμερα από ότι ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα τέτοιο μέλλον για την Ευρώπη και ε, επίσης όσον αφορά τους ε, Ευρωπαίους οι οποίοι είναι σαφώς πληρωτές όπως και η κυρία Μέρκελ η οποία λέει ότι αν έχουμε λιγότερα θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα θα μπορέσουμε να επενδύσουμε ε, για, αν δεν έχουμε λιγότερα θα μπορέσουμε να επενδύσουμε για να προχωρήσει η Ευρώπη και άλλοι έλεγαν όχι δεν δεχόμαστε να ε, επενδυθούν περισσότερα. Ε, δεν είχαν όλοι το ήρω όραμα που είχαν ε, στην εποχή τους ο Χέλμουτ Κόλ και ο Φρονσουά Μιτερό. Δεν θα ήταν η Ευρώπη σήμερα εκεί που είναι εάν δεν υπήρξαν αυτοί οι δύο ηγέτες και δεν θυμάστε ίσως πόσο κόστισε η επανένωση της Γερμανίας αλλά αυτό ήταν αναγκαίο για την υφή δεν μπορεί κανείς να προχωρά μόνο με κριτήρια οικονομικά και να λένε θέλουμε την Ευρώπη αλλά δεν πληρώνουμε για αυτήν. Δεν είναι παραδεκτό κάτι τέτοιο. Κύριε Βαν ε, μα είπατε για την ομιλία σας στο Συμβούλιο και ότι η κρίση δεν πάει χαμένη. Ε, δεν νομίζω το έλαβαν υπόψη τους όμως οι αρχηγοί κρατών, διότι εσείς και ο κύριος Γκαρόζο ήσασταν οι μόνοι οι οποίοι πραγματικά είχατε καλή εμφάνιση. Προ ε, τίνατε προϋπολογισμούς του οποίου δεν μου αρέσουν οι αριθμοί αλλά τουλάχιστον μιλήσατε για ανάπτυξη, για έρευνα, για προώθηση που είναι κάτι που χρειάζεται στην Ευρώπη και δυστυχώς οι αρχηγοί κρατών δεν το έλαβαν υπόψη ήθελαν να μειώσουν ε, τις πληρωμές τους και πρέπει να σας πω και στους δύο επιμείνετε, παραμείνετε σκληροί θα χρειαστεί ίσως ε, να κάνετε υπομονή και πιστεύω ότι είναι σωστή η θέση σας γιατί επιμείνατε, δεν υποχωρήσατε και γι' αυτό σας ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα ε, βρήκαν έναν αποδιοπομπαίο ε, τράγο τα μέσα ενημέρωση ότι ε, πέθανε η δημόσια διοίκηση ενώ είναι το 6% του προϋπολογισμού του συνολικού προϋπολογισμού λιγότερο από πόλεις σαν το Παρίσι ο στόχος μας ε, είναι όχι μόνο ε, δεν είναι να έχουμε τους καλύτερους θέλουμε αυτοί οι άριστοι να πάνε στην Παγκόσμια Τράπεζα ή σε ξένες ε, οργανώσεις και εταιρείες ε, εάν θέλουμε δηλαδή ε, να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε καλούς συναδέλφους, ε, χωρίς καλά στελέχη, δεν είναι δυνατόν να τους ζητάμε απαράδεκτες περικοπές. Όσον αφορά το Συμβούλιο, εδώ και 17 μήνες ξέρουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναμόρφωση της διοίκησης την οποία εκπώνησε το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την συζήτησε στην Επιτροπή και την ψήφισε χωρίς όμως να την σημειώσει καθόλου το Συμβούλιο να υπάρχει ένας τριμερής διάλογος διότι λαϊκίστικα παρουσιάζουν πρωτοφανείς προτάσεις αντί να διαπραγματευθούν συγκεκριμένα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελάτε στο Κοινοβούλιο Συμβούλιο, ελάτε στις επιτροπές μας να διαπραγματευτούμε για την αναμόρφωση της διοίκησης. Θα το πράξουμε και πρέπει να το ψάξουμε, αλλά δεν φτάνει να πληρώσουμε λιγότερα χρήματα, διότι δεν μπορεί η γραμμή να είναι less, less spending, much less spending, δηλαδή λιγότερες δαπάνες και αυτό να χαρακτηρίζει αυτό το Συμβούλιο. Και τελευταία παρατήρηση την ε, δεκάτη ε, του μηνός θα υπάρξει η απόδοση ενός βραβείου. Αλλά βλέπουμε ότι οι ίδιοι αρχηγοί κρατών που χρησιμοποιούν τους πόρους για την εξωτερική πολιτική, για την αναπτυξιακή πολιτική και θέλουν να τις περικόψουν αυτοί δεν αξίζει να λάβουν ε, το βραβείο Νόμπελ. Πρέπει να κερδίσουμε το βραβείο Νόμπελ, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με περικοπές στους διάφορους προϋπολογισμούς. Ας κάτσουν λοιπόν στα σπίτια τους αντί να πάνε στην απόδοση του βραβείου Νόμπελ και σκεφτούν πώς θέλουν να προχωρήσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα. Το λόγο τώρα ο κύριος Φερχόφστατ. Κύριε Πρόεδρε, ήταν αδύνατο, είπατε, να επιτευχθεί συμφωνία για τα 972 δις ευρώ. Μήπως ήταν καλύτερα να δούμε ετήσια τα ποσά, 139 δις, κάτι λιγότερο, ετησίως το 1 πεντηκοστό, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, του συνολικού προϋπολογισμού όλων των κρατών μελών της Ένωσης. 6,33 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός των κρατών μελών. Αυτό λοιπόν τελικά σημαίνει ότι αυτά τα 139 δις και το είπε και ο Ζωζεφ Ντόλ είναι 27 ευρώ κατά κεφαλή το χρόνο για τον κάθε πολίτη. Αυτό κοστίζει είναι γύρω στα 70 σέντ για τον καθένα από εμάς ε, την ημέρα. Και τι λέει ο κύριος Κάμερον, ότι αυτά τα 27 ευρώ ανά Ευρωπαίο πολίτη για όλο το χρόνο και τα 70 σέντ ημερησίως είναι πολλά και πρέπει να τα κατεβάσουμε γιατί τα 70 σέντ την ημέρα ανά πολίτη κατά κεφαλή είναι πάρα πολύ για τις χώρες αυτές. Εγώ το ξαναείπα και στο Στρασβούργο στην τελευταία συνεδρίαση, ε, αυτή τη συζήτηση θεωρώ παράλογη. Και είναι και ψέμα. Είναι ψέμα να λέει κανείς ότι οι περικοπές στον ε, προεπλογισμό της Ένωσης θα χρηματοδοτήσουν ε, ε, τις δημόσιες δαπάνες όχι, σε καμία περίπτωση. Μόνο με τη συγκέντρωση πόρων και τη συγκέντρωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατόν να μειωθούν δραστικά τα ελλείμματα στις χώρες μέλη. Και θα ήθελα να σας δώσω λίγα παραδείγματα γιατί έχουμε ε, στα εθνικά κράτη-μέλη διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων που εργάζονται παραδείγματο χάρη σε εθνικέ τράπεζε σε σχέση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στη ΣΥΠΑ ή γιατί στην Ευρώπη έχουμε διπλάσιου τριπλάσιου διπλωμάτε σε σχέση με τι ΗΠΑ. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε τριπλάσιου τετραπλάσιου στρατιώτε από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα γιατί να μην αντικαταστήσουμε επενδυτικά προγράμματα στην έρευνα, στην ανάπτυξη, υποδομές, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση μέσω των ομολόγων έργων, των project bonds. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, συγκεντρώνοντα πόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όχι να τσακωνόμαστε για 70 σέντ, 79 σέντ την ημέρα. Αυτό που πρέπει να πετύχουμε σήμερα είναι να συμφωνήσουμε στο τι μπορούμε να συγκεντρώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να μειωθούν και τα κρατικά ελλείμματα. Και νομίζω ότι είναι μια καλύτερη άσκηση από αυτή που κάνουμε σήμερα, δηλαδή ε, μελλοντικές υποδομές, ανάπτυξη, έρευνα, περικόπτονται οι σχετικές δαπάνες. Τι άλλο περικόπτεται και το μέλλον ουσιαστικά της Ευρώπης. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το, τελικό, το τελευταίο νούμερο, ε, το τελικό συγγνώμη νούμερο. Δύσκολο κανείς να το μαντέψει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι στο τέλος θα υπάρξει συμφωνία. Και εγώ νομίζω ότι θα γίνει όπως έγινε και πριν από έξι χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς κύριε Φων Ρομπέη, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είπατε ότι δεν πήρε και το βραβείο Καλιστίων ε, ο προπολογισμό εκείνη τη ε, χρονιά, ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι εντάξει, μπορούμε να δώσουμε λίγο λιγότερα σε κάποιε χώρε, λίγο παραπάνω σε κάποιε άλλε, λίγο περισσότερε επιδοτήσει σε κάποιε τρίτε χώρε. Και τελικά θα κάνουμε τα ίδια με αυτά που κάναμε το 2006. Με 30-40 παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις για να μπορέσουμε να τις εξαγοράσουμε όλους τελικά σαν ένα jackpot που όμως το κερδίζουν όλοι ή τα αερομιλιών. Έχουν αερομιλιών ε, οι πολίτες, αερομπιλιών όμως οι ε, χώρες μέλη της Είναι ένα παιχνίδι. Πώς θα το σταματήσουμε αυτό. Πρέπει να σταματήσουμε τις εισφορές τις εθνικές. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο χρηματοδότησης της Ένωσης. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Και γι' αυτό ελπίζω ότι αυτό το κεφάλαιο για την εισαγωγή, δηλαδή πραγματικών ιδιών πόρων, ελπίζω να το διατηρήσετε αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, ο προπολογισμό να ε, μην βασίζεται στι εθνικέ φορέ, γιατί αυτό σκοτώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αν στηρίζεται σε ίδιου πόρου, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι σημαντικότερο το ευρωπαϊκό από τα εθνικά συμφέροντα και σα παρακαλώ κύριε Φωνρομπέη να διατηρήσετε ανοιχτό το κεφάλαιο αυτό, να έχουμε το φόρο για τι χρηματοπιστωτικές συναλλαγέ. να έχουμε τον ΦΠΑ το 2021 ω νέο ίδιο πόρο, ώστε αυτό το παιχνίδι που βλέπουμε σήμερα να παίζει να σταματήσει πια. Και μπορώ να σα πω, είναι, ξα... είναι ξεκάθαρη θέση του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου, το είπε ο πρόεδρος Ζωζεφ Ντόλ, ήδη οι πόροι. Και κατάρρισε αυτής της ε, που υπάρχει Αλλιώς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόφστατ. Κύριος Κον Μπεντίτ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, για να συνεχίσω μετά από αυτά τα οποία είπε ο Γκί, πιστεύω ότι σήμερα βρισκόμαστε το τέλο ενό προτύπου πολιετών προπελών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε 27, δεν είμαστε 28, είμαστε 29. Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το ίδιο δικαίωμα αρνησικυρία με του άλλου 28. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λησμονούμε πολύ συχνά στι διαπραγματεύσει. και κυρίω αυτέ που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτό. Διότι πιστεύω ότι οι αρχηγοί κρατών είναι κάπω σαν του γονεί Μα λένε ακούστε παιδιά, μια φορά όταν θα αρχίσουμε λίγο να τους ε, κάνουμε μάθημα και τους κάνουν τι θέλουμε θα μας ακούσουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ελπίζω ότι έχει ενηλικιωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα είναι ενεργή, δεν θα ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο λέξα για τους ιδίους πόρους, είναι προφανές ότι η καλύτερη λύση για να σταματήσει αυτού του είδους το τσίρκο είναι να σταματήσει αυτού του είδους η Ευρώπη και να μειωθούν οι εθνικές συνεισφορές. Ναι, είμαστε υπέρ των να μην πληρώνουν τίποτε από τον εθνικό του προϋπολογισμό τα κράτη-μέλη. Έτσι θα έχουν το δικό τους εθνικό προπολογισμό και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η καινοτομία την οποία θέλουμε να κάνουμε. Ελέγχθηκε αυτό. Και αυτό είναι προφανές. Κάτι άλλο όμως με εκνευρίζει σε αυτή τη συζήτηση. Ας πάρουμε τη Γεωργία. Όλοι θέλουν να μειωθούν οι δαπάνες. Αλλά όταν γίνονται οι προτάσεις για ανώτατο όριο σε 300, από 300 σε 100 εκατομμύρια ευρώ, αυτά τα οποία δίδονται σε μία γεωρική δραστηριότητα, ποιες χώρες λένε όχι, ποια είναι η πρώτη χώρα που λέει όχι. Η Αγγλία, για την αυτού μεγαλειότητα τη βασίλισσα της Αγγλίας λέμε όχι. Και αυτό ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση της Αλληλεγγύης. Ναι, πρέπει να επανορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμονται τα κονδύλια. Και στη Γεωργία, αν έχουμε ανώτατο όριο 100 εκατομμύρια ευρώ, διότι ξέρουμε ότι 70% της βοήθειας στη Γεωργία δεν είναι περισσότερο από 18 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ανώτατο όριο 300 εκατομμύριων ευρώ για κάποιου και η Γερμανία και η Αγγλία είναι οι πρώτε χώρε που λένε όχι σε αυτό το ανώτατο όριο. Θα κανονίσουμε έτσι 7 δι τα οποία θα μπορούσαμε να επανεπενδύσουμε στην ε, κατανομή πόρων για τις υπαίθριες ζώνες που τι οποίε θέλουμε να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Και αν το θέλουμε να το κάνουμε αυτό, έτσι θα πρέπει να ενεργήσουμε. Θα σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Είπατε ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν μπορεί να είναι προπολογισμό αντικυκλικό. Ναι, αυτό είναι και εν μέρει αληθέ και εν μέρει ψευδέ. Διότι εάν ε, μπορέσουμε ε, για κάποιες περιπτώσεις να προβλέψουμε κάποια κονδύλια έχουμε να κάνουμε αντικυκλικό. Δεν είναι όμως προφανές αυτό για όλους, αλλά για κάποιες περιοχές αυτό είναι δυνατόν. Σήμερα, λοιπόν, η ευφυΐα μας να μπορέσουμε να στοχεύσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις θα αποτελέσει την προστέμενη αξία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και μας λένε ναι, ναι, ναι, αλλά θα πρέπει να μάθει να δαπανεί καλύτερα τα χτήματά της η Ευρώπη. Κοιτάξτε, κοιτάξτε όλα τα ελεκτικά συνέδρια της ε, Ευρώπης, όλοι κάνουν παράλογε δαπάνε. 70% του χρήματο το οποίο δαπανάτε από την Ευρώπη δαπανάτε ετήσι των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για αυτή την τρέλα, αλλά δεν έχουν το θάρρο να πούν εμείς είμαστε ανεύθυνοι, γι' αυτό στρέφουν το δάκτυλο προς τις Βρυξέλλες και στα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όμως έτσι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, δεδομένου ότι και ο Ευρωπαϊκό ΦΠΑ είναι ένα άλλο θέμα. Σήμερα κατανοήσαμε ότι χρειαζόμαστε κοινοτικό προπολογισμό και 1% του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι το ΑΕΠ. Το 1932 όταν τα Ευρω... ΗΠΑ έκαναν τον νομοσπονδιακό τους προπολογισμό ήταν στο 1% και σήμερα εκεί βρισκόμαστε. Το 42 ήταν το 100% του ΑΕΠ σήμερα είναι το 23% του ΑΕΠ του Αμερικανικού. Αυτοί όμως που θέλουν ε, ενωμένη Ευρώπη, ομόσπονδο Ευρώπη, πρέπει να παρέχουν τα μέσα σε αυτή την Ευρώπη να ενεργεί η όφελος των Ευρωπαίων. Εάν δεν τις δώσουμε τα μέσα, θα πούνε οι Ευρωπαίοι πολίτες σε τι μας χρησιμεύει η Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν τους πολίτες τους. Το βλέπουμε αυτό στις κρίσεις. Και θα ήθελα τώρα να πω κάτι για αυτό το οποίο συμβαίνει την παράλληλη κατάσταση της Ελλάδας. Ναι ή όχι καταλάβαμε όλοι ότι σήμερα θα πρέπει να υπάρχει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους διότι δεν μπορούν να την ε, οι Έλληνες. Και όσο περισσότερο περιμένουμε, όσο περισσότερο επιδένουν την κατάσταση διότι δεν χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέσα. Και τι κάνουμε, δίδουμε χρήματα στους επενδυτές εκτός Ευρώπης. Παίρνουμε χρήματα από τους Ευρωπαίους πολίτες για να πληρώσουμε επιτόκια σε αυτούς που βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Εφιέστατο είναι αυτό, ποτέ δεν είχα δει κάτι τόσο εφιές. Για να τελειώσω λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ο προπολογισμό βάσει της πρόταση της Επιτροπής είναι το μίνιμουμ, το ελάχιστο. Εάν κατέβουμε χαμηλότερα, εμείς θα πούμε όχι, δεν θα πρόκειται σε αυτή την περίπτωση για προϋπολογισμό για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ όλους τους ομιλητές να σέβονται το χρόνο τον οποίο έχουν. Το χρόνο τώρα έχει ο κύριος Τσαραντήλ για δυόμιση λεπτά. Το πολύ κύριε Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και πρέπει να σας πω ότι παρότι είμαι μέλος του θεσμικού αυτού οργάνου, δεν θεωρώ ότι είναι πάντοτε αναγκαίο να αγωνιστώ με αυτό και για αυτό, ιδίω σε περιπτώσεις όπου το μόνο που κάνει είναι να ε, παλεύει κατά των άλλων θεσμικών οργάνων ουσιαστικά μόνο και μόνο για την ιστεροφημία του ή για την καλή του φήμη. Αυτό συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ε, ουσιαστικά μια παράσταση για το Θεαθήνη, για, το, ε, για τους λαούς της Τίποτε ε, περισσότερο. Καμία εθνική κυβέρνηση δεν είναι αντίπαλος ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κατ' κάθε εθνική κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι εταίροι. Είναι εταίροι στους πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Γι' αυτό και είμαι πολύ κατά όλης αυτής τη ρητορία της πολεμικής με τη... για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ολοκληρώστε ο Ρεκονπεντήτ. Μάλιστα. Ωραία. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι το μέγεθος του προπολογισμού, αλλά η δομή του προπολογισμού. Αυτό έχει σημασία. Και πιστεύω ότι εμείς και εσείς κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να δείτε πιο προσεκτικά τη δομή του προπολογισμού που είναι ο πυρήνας, είναι το κεντρικό ε, σημείο. Δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε αποτυχία, αλλά κάτι πολύ απλό βλέπουμε. Ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κυβερνήσεων που θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ζει ε, με τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Ούτε μπορούμε να κατηγορούμε πάντοτε τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες κυβερνήσεις και άλλοι πρωθυπουργοί και άλλοι καγκελάροι που τοποθετήθηκαν ε, με παρόμοιο τρόπο κυρία Μέρκελ από το ΕΛΚ, κύριο Φερχόφστατ, ε, ε, να του μάλλον φιλελεύθερη, ε, να πω στον κύριο τα λοιπά. Επομένως, το πρόβλημα είναι γενικότερο. Σας παρακαλώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, θερμά σας παρακαλώ, να μην δείτε μόνο τις κατηγορίες του περιπολογισμού όταν λαμβάνετε τις αποφάσεις σας. Για να έχουμε συμφωνία που θα μπορεί να είναι αποδεκτή από όλου θα πρέπει να την πετύχουμε μόνο με τον εξή τρόπο. Με αναλυτική εξέταση του προπολογισμού που θα δει τι αποτελεί προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι δεν αποτελεί. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας. Τώρα, σε ό,τι του ίδιου πόρου. Και είναι η τελευταία μου παρατήρηση. Υπάρχει ιδεολογική συζήτηση. Οι μεν που θέλουν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, οι άλλοι θέλουν το... Και, το Ευρωπαϊκό Υπεκράτο και άλλοι δεν το θέλουν. Αυτοί που θέλουν το υπερκράτο φυσικά και θέλουν ε, και του ίδιου πόρου. Αυτοί που δεν το θέλουν δεν θέλουν του ίδιου πόρου. Και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή δεν είναι ομοσπονδία, ποτέ δεν θα γίνει ομοσπονδία. Σα παρακαλώ λοιπόν μην ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω να σέβεστε το χρόνο. Σας παρακαλώ για να μπορέσουμε να καλύψουμε ε, όλους αυτούς που θέλουν να μιλήσουν. Το λόγο έχει, ζητάει η κυρία Ανδρέασεν. Πρόεδρε, δεν είστε κύρια Μέρκελ, γι' αυτό δεν θα σας ζητήσω να πείτε στον Κάμερο να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Νάιτζελ Φάρε το έχει καταλάβει πάρα καλά, αλλά δεν είπε στον Κάμερον η Μέρκελ να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να το, να το σκεφτόμαστε όταν διαπραγματευόμαστε για τον προπολογισμό. Δεν εκπλήσω που δεν υπήρξε συμφωνία και υπήρχε αποτυχία στι διαπραγματεύσει την προηγούμενη εβδομάδα. Σε περίοδο κρίση, περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι θέλουν να είναι αποδοτικέ οι επενδύσει του. Η ατζέντα τη ε, Λισαβόνα που ε, τιολογεί το παρόντα ε, πλαίσιο δημοσιονομικού πλαισίου είναι αποτυχία. Όλα τα χρήματα απέτυχαν και σήμερα αντί να έχουμε την ε, ανάπτυξη που μας είχαν υποσχεθεί έχουμε στασιμότητα. Αντί να έχουμε θέσει απασχόληση, έχουμε ανεργία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι δεν ε, θέλουν να απομισθούν την ευθύνη του στα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα. Αλλά πρόκειται για πολιτικέ που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κονταϊλιά τα οποία θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει που δημιούργησε αυτή την κατάσταση για δέκατη συνεχή χρονιά το ελεκτικό συνέδριο δεν θέλησε να χορηγήσει την απαλλαγή και είπε ότι δεν πήγε στα σωστά άτομα για τους σωστούς, ε, σωστές πολιτικές το χρήμα. Έχουμε μεγάλο ποσοστό σφάλματος και όλοι θα πούνε ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα. Βεβαίως τα προγράμματα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που θα πρέπει να σταματήσει το χρήμα το να πηγαίνει στα κράτη-μέλη που παραβιάζει τους κανόνες. Θα πρέπει να το κάνει και ζητάτε περισσότερα χρήματα χρήματα για αυτές τις χώρες που τα σπαταλούν τα χρήματα. Υπάρχει λογική σε αυτό. Στην πραγματικότητα, ο προϋπολογισμός και το πλαίσιο δημοσιονομικού πλαισίου ήταν πάντα κάτι το δύσκολο. Όλο και περισσότερο χρήματα ζητούνται για σχέδια τα οποία δεν έχουν νόημα. Δόθηκαν στα διαθετικά ταμεία στην Ισπανία 130 δις τι έκανε. Τι έκανε η Ελλάδα με τα 60 δις για τα διαρθρωτικά της ταμεία. Νομίζω ότι πήγατε σε αυτή την ε, διαπραγμάτευση χωρίς ε, να υπάρχει συμφωνία για το προβλήμα του 2013, παρά το γεγονός ότι είχαμε συμφωνήσει για τον διαθωτικό προπλησμό του 2012. Τα αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων νομίζετε ότι είναι ανόητοι και θα συμφωνήσουν με αύξηση 2,7 και διορθωτικό το Σεπτέμβριο 7% ως αύξηση. Πρέπει να γίνουν επιλογές. Αυτό είναι το θέμα. Επιλογές. Εάν μιλούμε για αλληλεγγύη, πράγμα το οποίο θα, θα πρέπει να αναφέρουμε, αλλά να μιλούμε περισσότερο για επικουρικότητα, θα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Δεν χρειαζόμαστε την υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής ούτε την υπηρεσία όπως είναι με την ιστορία της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ζήμερ. Το Κοινοβούλιο πριν από τις διαπραγματεύσεις είπε σαφώς ότι υπάρχει μία κόκκινη γραμμή για το Κοινοβούλιο και η πρόταση του κυρίου Βαν Ρομπόι δεν είναι αποδεκτή για μας. Και η πράσινη και η αριστερά είπαν ότι η απόλυτη γραμμή, η κόκκινη γραμμή είναι αυτή, δηλαδή η πρόταση της Επιτροπής. Πρέπει να σας πω ότι στην πρότασή σας πολλά δεν έχουν ρυθμιστεί, διότι το ποσό το οποίο είναι αμφιλεγόμενο είναι το 0,01% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τσακώνονται για το τίποτα. Ενώ το ερώτημα είναι πού πηγαίνει δημοσιονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος θα πρέπει να εξασκεί την επιρροή στο μέλλον. Είναι ε, η πολιτική των διαρθρωτικών ταμείων, των εκπτώσεων, ποιος δηλαδή ε, έχει εκπτώσεις και ποιος πληρώνει τις εκπτώσεις αυτές. Δηλαδή ε, ποιος ωφελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος ισοπεδώνεται και όπως και στην προηγούμενη διάσκεψη κορυφής νομίζω ότι ένα σωρό ερωτήματα μείναν αναπάντητα. Τι θα γίνουν στις δύο-τρεις επόμενες εβδομάδες μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Ε, τα βασικά δεν θα αλλάξουν. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι θα πρέπει στο τέλος να πούν εμείς τι αποκομίζουμε. Κάθε εθνική κυβέρνηση η οποία κάνει τέτοια διαχείριση οικονομική θα είχε εκδιωχτεί. Και εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουμε την πορεία μας χωρίς να λέμε ότι σαν, ε, Ευρωπαϊ... Ε, σαν Ευρωβουλευτές είμαστε υπόλογοι στις χώρες μας και πρέπει να εξηγήσουμε γιατί παρουσιάζουμε αυτές τις θέσεις. Τουλάχιστον η... στη Γερμανία η γερμανική αριστερά και υποθέτω και άλλοι συνάδελφοι θα πρέπει να μπορέσουν να επηρεάσουμε τη διαμόρφωση της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε Βαν Ρόμποη, αυτές τις εβδομάδες αποφασίζετε τι θέση εσείς θα έχετε στην ιστορία και ε, πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα είστε, θα ε, μία μαριονέτα, ένας μάγος ή μαγεμένος. Διότι εδώ βλέπουμε ότι ε, υπάρχει μία άποψη που αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε είμαστε σε κρίση. Πρέπει να ε, λύσουμε το πρόβλημα του ελλείμματος δημοκρατίας και ε, το σκιάχτρο ενός παγκοσμίου πολέμου. Μακάρι να μπορούσατε να γίνετε μάγος, να καταλάβετε ότι υπάρχουν τόσο πολλές ανησυχίες ε, τις οποίες εκδηλώνουν οι πολίτες ε, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι καθοδόν μεν αλλά ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών μεγαλύτερη ε, συναπόφαση και θα πρέπει να ζητήσετε να υπάρχει μία συνέλευση η οποία θα μπορέσει να επιλύσει αυτά τα προβλήματα και αυτό όντως θα γίνει μόνο εάν μπορέσουμε να κάνουμε μία μεγάλη ανακατανομή την πιο μεγάλη που έχει γίνει εκτός πολεμικής περίοδου ε, δηλαδή είναι μία ανακατανομή η οποία έχει γίνει από τις χρηματαγορές που εκπροσωπούν εδώ ο κύριος Φαράζ και η, η ε, πολιτική του ομάδα για τα 22 δισεκατομμύρια τα οποία κρύπτονται ε, σε σκιώδεις τράπεζες. Εάν λοιπόν μπορέσετε να σταματήσετε αυτό το παγκόσμιο πόλεμο ε, και να προχωρήσετε τότε θα μπορέσουμε να έχουμε και μία ανάπτυξη πέραν του 0,3%. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Λαμασούρ, πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, από την Ευρώπη των 12, χαμογελώντας, Λέγαμε ότι είχαμε 11 ευθύνοντε στο τραπέζι που μιλούσαν για την Ευρώπη και την κυρία Θάτσερ που μίλαγε για τα λεφτά τη. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε 27 κυρίε Θάτσερ να συζητούν. Και το μόνο που συζητήτων ήταν περικοπέ, περικοπέ, περικοπέ. Όλοι είναι τυφλοί και όλοι θέλουν να σώσουν τη δική τους παρτίδα, χωρίς να καταλαβαίνω ότι τελικά κόβουν τον κορμό, άρα όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία προτείνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα χαιρετούμε και την Ατζέντα 2020 και το Σύμβολο για την Ανάπτυξη και την Ευρώπη ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή. Και πρέπει να προσέξει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να είναι αξιόπιστο. Πώς μπορούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να λένε ότι αποφασίζουν για το προπολογισμό τη Ένωση μέχρι το 2020, αν δεν μπορούν ούτε καν να εκτελέσουν το προπολογισμό του 2012 μέσω των αρμοδίων υπουργών τους η κατάσταση όπως την επενθύμησε ο πρόεδρος Μπαρόζο, αλλά έχουμε και χειρότερα ακόμα. Ο Ευρωπαϊκός Περιπολεγισμός είναι ήδη ο μικρότερος κοινό παρονομαστής. Έχει γίνει αυτό που μας χωρίζει περισσότερο, ο πιο μεγάλος διαιρέτης αν θέλετε, διότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εντάσεις λόγω της κρίσης και έχουμε και ένα σύστημα που θέτει αντιμέτωπες τις 12 χώρες που συνεισφέρουν και τις 12 χώρες που είναι δικαιούχοι, μια κατάσταση που είναι απαράδεκτη πλέον για τους φορολογουμένους των πρώτων χωρών, αλλά και ταπεινωτική κατάσταση για τους ε, πολίτες των δεύτερων χωρών. Και είδαμε ότι πήγε η Άγγελα Μέρκελ ε, στη Λισαβόνα, πήγε στην Αθήνα. Αυτές οι αναταρχές που είδαμε εκεί είναι μια προειδοποίηση. Η Ευρώπη μπορεί να συμφιλιώσει λαούς, αλλά μπορεί να γίνει και ένα εργαλείο που τελικά ε, θα τους φέρει αντιμέτωπους τους μεν προς τους δε. Τέσσερα κλειδιά έχουμε για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο όμω. Το πρώτο το είπατε μόνο σα, ε, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να επανέλθουμε στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Ναι, για το rebate των Βρετανών. Όχι να το μειώσουμε, να το αυξήσουμε και για το γερμανικό rebate και να βάλουμε και άλλες χώρες μέσα ε, και να ξεκινήσουμε τους δικούς μας ίδιους πόρους. Δεύτερο κλειδί το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολισμό για να δαπανίσουμε καλύτερα τους πόρους στις Βρυξέλλες. Και αυτό τι θα πει, θα πρέπει και την αμοιβεοποίηση, τη συλλογική διαχείριση να την αξιοποιήσουμε, ώστε ο καθένας στις χώρες τους να δαπανά λιγότερα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αφεύρει. Ας το χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το σκοπό. Τρίτο κλειδί, συνοχή μεταξύ χρηματοοικονομικής αλληλεγγύης και δημοσιονομικής αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είδε διαφορετικά τα δύο θέματα λάθος, διότι είναι οι δύο του ίδιου νομίσματος. Ε, θα πρέπει η δημοσιομική ικανότητα να θεωρηθεί μιας, ως μια νέα προσέγγιση του ε, προϋπολογισμού και όχι ως εναλλακτική λύση. Και ολοκληρώνουμε το τέταρτο κλειδί, κύριε Πρόεδρε, ρήτρα της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Να είμαστε ρεαλιστές και μετριοπαθείς, ε, ταπεινόφρονες. Κανένας μας δεν μπορεί να ξέρει τι θα φέρει συγκυρία για την κάθε χώρα του χρόνου. Η εντολή του Ευρωκοινοβουλίου εκπνέει σε 18 μήνες. Ε, το πολιτές ε, λοιπόν γνωσιαμικό σχέσιο θα ολοκληρωθεί όσο θα έχουμε το κοινοβούλιο ε, που θα έχει εκλεγεί, δηλαδή το 2019. Άρα πρέπει να δώσουμε στους διαδόχους μας και στους διαδόχους των διαδόχων μας τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να πετύχουν. Ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ κύριε Λαμασούρ. Νομίζω ότι παρουσιάστε μία πολύ σαφή και πλειοψηφική ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα για τις απαντήσεις ξεκινάμε τον κύριο Μπαρόζο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συμφωνώ διότι θέλω να ε, παρουσιάσω και να διασκεδάσω τις ανησυχίες των ε, άλλων ομιλητών, τις οποίες συμμερίζομαι. Ήθελα να πω δύο λόγια. Όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πολλές ώρες υπομονητικά ήμουν και εγώ εκεί, με υπομονή και είδα πώς διεξήθηκαν τα... Αλλά το καθήκον του Προέδρου είναι να μπορέσει να καταλήξει συνένεση, συμβαστική λύση μεταξύ των κρατών μελών. Και ξέρετε σήμερα πόσο αυτό το εγχείρημα είναι δύσκολο. Κατά διάρκεια των συζητήσεων είχα την δυνατότητα, δεδομένου ότι κάποιοι μίλησαν για τις συζητήσεις οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν, να ανατρέξω στην δική μου εμπειρία. Ήμουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύο φορές ήδη σε αυτή την κατάσταση. Το 1992 Ω υπουργό Εξωτερικών τη χώρα μου συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο ενέκρινε τις ε, δημοσιονομικέ προοπτικέ. και τότε ο πρόεδρος του Συμβουλίου ήταν ο κύριος Μέιτζερ Είχαμε τότε τον κύριο Μιτερό, τον κύριο Κολ και άλλους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων ήμουν παρόν. Και με την Βρετανική Προεδρία έγινε πάρα πολύ σημαντική αύξηση των πόρων της Ευρώπης. Μετά, ως πρόεδρος Επιτροπής συμμετείχα στην ε, κατάρτιση του προπολογισμού και στις συζητήσεις που έγιναν για το 2005. Ο Τόνι Μπλέαρ του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν προεδρεύων και παρόλα αυτά έγινε πάλι σημαντική αύξηση των πόρων που διατέθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα λοιπόν, τι καθιστά τόσο δύσκολη την δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας. Έθεσα το ερώτημα στους αργούς κατών κυβερνήσεων και το θέτω και σε εσάς. Και η παρατήρηση μου είναι η εξή. Για πρώτη φορά, ίσω εξαιτία τη παρούση οικονομική κρίση, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση στην οποία συζητούμε κυρίω περικοπές για τον προπολογισμό. Και όντω υπάρχουν κάποιε κυβερνήσεις που δεν είναι ικανές να παρουσιάσουν στην κοινή τους γνώμη μια θετική εικόνα για την ε, Ευρώπη. Ακόμη και η κυρία Θάτσερ, την οποία ανέφεραν κάποια από εσά, θα πω ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας είχαμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον προσμό. Βεβαίως το τίμημα που πλήρωσαν οι άλλες χώρες ήταν η περίφημη επιταγή που δόθηκε, το τσεκ που δόθηκε στους Άγγλους. Αλλά με την κυρία Θάτσερ, επαναλαμβάνω, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των πόρων του κοινοτικού προπολογισμού. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα και αιτιολογείται αυτή η κατάσταση. Όντως, δεν είμαστε πάντα σε εθνικό επίπεδο σε θέση να εξηγήσουμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα ευρωπαϊκά μέσα για την πολιτική μας. Και βεβαίως δεν μπορώ να δεχθώ κάποιες δηλώσεις όπως αυτές που έγιναν σήμερα και αναφέρονται στο ότι δεν χρειαζόμαστε την κοινή εξωτερική υπηρεσία. Συγγνώμη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενέκριναν την συνθήκη που την ε, δημιούργησε. Είναι υποχρεωμένε λοιπόν να σεβαστούν τι δεσμεύσει και την υπογραφή του. Βεβαίω, μπορούμε να διαφωνήσουμε με τα ποσά. Αλλά πολλέ φορέ υπάρχει και πρόβλημα ιδεολογικό. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν όλα τα να αναγάγουν σε ιδεολογία. Με αρνητική μνήα για την Ευρώπη, λέγοντα ότι ο αποδιοπομπαίο τράγο για την κρίση είναι η Ευρώπη. Ενώ είναι η απάντηση για την επίλυση τη κρίση η Ευρώπη. Και βεβαίω έγιναν κάποιες δηλώσεις ε, για έλλειμμα αποδοτικότητας ε, της Ευρώπης, αλλά πού καταλήγουμε εκεί. Θέλουμε λιγότερη Ευρώπη. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό εξηγεί και την αντίφαση την οποία εξέφρασε ο κύριος Κομπεντίτ. Δηλαδή, ζητούμε συγχρόνως μείωση των δαπανών των αγροτικών και η ίδια αντιπροσωπεία είναι κατά της πρώτας επιτροπής που συνίσταται στην χορήγηση ανωτάτου ορίου ε, για τις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό είναι παράλογο και θα μπορούσα να παραθέσω και πολλά άλλα παραδείγματα τέτοιων αντιφάσεων. Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας κ. Σβόποντα είπε ποιος πρόσφυσε τα συμφέροντα της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων και η Ευρώπη θα μπορούσα να σας πω κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων. Το είπαμε με απόλυτη σαφήνεια και αποφασιστικότητα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Σούλτ, στην αρχή επίσης έκανε μια παρέμβαση ε, φιλόδοξη, αλλά μπορώ να πω με ανοιχτό πνεύμα για επίτευξη συνενετικών λύσεων, διότι πρέπει μεταξύ όλων ημών να καταλήξουμε σε συνενετική λύση. Και για να είμαι δίκαιο, πρέπει να πω ότι και πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επέδειξαν επικοδομητική στάση. Κάποιοι είπαν ότι εν μέσω αυτή τη συζήτηση μεταξύ των ε, συνεισφερόντων καθαρά και αυτών που δικαιούνται ε, τα ποσά, υπάρχει πρόβλημα. Και το είπε και ο κύριος Λαμασούρ. Πράγμα το οποίο πολλές φορές θέτει ένα αμφιβόλο και την βασική αρχή της αλληλεγγύης. Είπε κάποιος ότι όλοι είμαστε καθαροί, θετικοί δικαιούχοι, αποδέκτες των πόρων της Ευρώπης, γιατί είναι κοινό σχέδιο όλων μας η Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, κάνοντας κάποιες συγκρίσεις, τι είδα, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο με τον προϋπολογισμό για την έρευνα κέρδισε πολύ περισσότερο στο προϋπολογισμό 2007-2013 στα πλαίσια των προγραμμάτων τα οποία υποφελείται από πολλές άλλες χώρες που είναι στα πλαίσια τη συνοχής. Είναι λοιπόν μύθος αυτό που επικρατεί στην Ευρώπη. Ότι δηλαδή όλα τα χρήματα πηγαίνουν στι φτωχέ χώρες, στις χώρες της συνοχή. Οι χώρες, οι net contributors, οι καθαροί εισφορεί επίση επωφελούνται πάρα πολύ από τα κοινά κοινοτικά προγράμματα. Και μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν και προευρωπαϊκά πολλά μηνύματα γύρω από την τράπεζα. Πρώτα απ' όλα το θέμα της ομοφωνίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, ο οποίο προσπάθησε να διατηρήσει την ισορροπία της πρότασης τη Επιτροπής. Και βεβαίω εδώ συμμερίζομαι τι ανησυχίε του κυρίου Φέρχοφστατ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι ω το τέλος, διότι όντω οι πιέσει οι οποίε προέρχονται πολλέ φορέ από κάποιε πρωτεύουσε και πρέπει να σα πω ότι αυτό το είδαμε μεγάλη μου λύπη, δεν είναι η ουσία δεν είναι μόνο τα ποσά, αλλά θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι κανένας άλλος δεν θα πάρει τόσα πολλά ή ότι οι άλλοι θα δώσουν περισσότερα κονδύλια. Είδα μια αντιπροσωπεία την οποία ενδιαφέρει περισσότερο να ξέρει πόσο πληρώνουν οι άλλοι και πόσα παίρνουν παρά να ενδιαφερθούν με τα δικά τους ποσά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί, διότι αποδεικνύει ότι όντως χρειαζόμαστε μεταξύ όλων ημών που είμαστε υπεύθυνοι για την Ευρώπη να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους Ευρωπαίους. Θα σας αναφέρω και ένα σχόλιο ενδιαφέρον από κάποιο Πρωθυπουργό. Τι είπε. Αυτό που λέτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι σημαντικό. Διότι κάποιοι από εμά υπενθυμίσαμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ο πρόεδρο σα το είχε κάνει, αλλά και εγώ επίση, καθώ και άλλε αντιπροσωπείε. Και είπαν κάποιοι, πώ είναι δυνατόν ή τα ίδια πολιτικά κόμματα να λένε άλλα μέσα των πολιτικών της ομάδας του Ευρωπολίγα, αλλά εδώ σε επίπεδο αρχών κρατών και κυβερνήσεων. Προσέξτε το αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό. Οι πολιτικές ομάδες, οι οποίοι είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής και σας ευχαριστώ, διότι θα πρέπει να προσέξετε ώστε και τα κόμματά σας σε εθνικό επίπεδο να λένε τα ίδια πράγματα. Ξέρω ότι είμαστε από διαφορετικέ πολιτικέ οικογένειε, αλλά δεν θυμάμαι και ότι εντό τη ίδια πολιτική οικογένεια πολλέ φορέ είναι προφανή τα πράγματα για όλου εμά που θέλουμε να έχουμε μια πιο αλληλέγγυα Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να σα αναφέρω. Επίση πρέπει να προσθέσω το εξή. Δεν θα πρέπει να δεχθούμε αυτέ τι λαϊκίστικε επιθέσει, οι οποίε είναι υπεραπλουστευμένε και αρνητικέ για τον κοινοτικό προβλησμό. Βεβαίω υπάρχουν σφάλεσμα και πολλέ φορέ ε, αναφέρονται κάποια περί απάτης. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κυρία Ντρέισεν, ξέρω ότι πολλές φορές πρόκειται για σφάλματα που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο, αλλά μην νομίζω ότι η Κομισιό δεν κάνει τίποτα. Πολλές φορές τα κονδύλια σταματούν να τρέχουν προς αυτές τις χώρες. Στην Τσεχία έχουμε σοβαρά προβλήματα ε, διαφθοράς εξαιτίας του συστήματος που υπάρχει στην περίπτωση της Τσεχίας σταμάτησαν να τρέχουν τα κονδύλια για τη χώρα αυτή. Είναι έτοιμη λοιπόν να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν εντοπίσει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Βεβαίως, όχι βάσει ε, συγκεκριμένων στοιχείων, αλλά βάσει συγκεκριμένων εκθέσεων. Αυτό το λέγω για να προσπιστώ τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό και να μιλήσω για την συνοχή. Και υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο συλλομώ. Είναι αληθές βεβαίως ότι τα κοινοτικά ε, ταμεία με τα κονδύλια που χρήσαμε δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει να κάνουμε και τη δική μας αυτοκριτική. Κάποια προγράμματα όντως δεν κατέληξαν πάντα στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γι' αυτό στα πλαίσια των προτάσεων για την μελλοντική φάση είπαμε ότι θα πρέπει τα προγράμματα να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων που έχουμε ε, σχεδιάσει από κοινού. Στα πλαίσια κυρίως της Ευρώπης 2020. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν μπορεί κανείς ε, ε, να χορηγεί κονδύλια και να μην κάνει επίκριση, ανάλυση και εξέταση όλων των δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι θα το κάνουμε βεβαίως για να βελτιστοποιήσουμε την χορήγηση των κονδυλίων για να ελέγξουμε τι ακριβώς γίνεται και για να έχουμε καλύτερο το ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Αλλά δεν θέλω με αντιευρωπαϊκά ε, λαϊκίστικα σχόλια για τον κοινοτικό προπολογισμό που είναι μια επίθεση στα θεσμικά όργανα και στους Ευρωπαίους αξιωματικούς να συμφωνήσω. Γι' αυτό συνεχίζω να σκέφτομαι ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμβαστική λύση. Θα πρέπει σε αυτή τη φάση να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην πάρα πολύ δύσκολη αναζήτηση τέτοιου είδου λύσεων, αλλά συγχρόνω θα πρέπει να απαιτήσουμε από όλε τι κυβερνήσει να κάνουν σοβαρή συζήτηση. Και θα ήθελα να υπολογίσω στην σοβαρότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξηγήσουν με απόλυτη σαφήνεια, όχι μόνο εδώ και στο Στρασβούργο ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε, σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε, γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε έναν προπολογισμό για την ανάπτυξη τη Ευρώπη. Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν θα καταλάβουν ότι εν μέσω μια τόσο σοβαρή οικονομική κρίση από την απαρχή τη δημιουργία Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται περικοπέ και δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην αηφόρο ανάπτυξη, στην κοινωνική ε, ανάπτυξη που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους πολίτες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε Μπαρόζο. Ο Πρόεδρος Βαν Ρομπάι τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους παρατήρησαν και συνειδητοποίησαν ότι προασπίστηκα έναν προπολογισμό που παρά το γεγονός ότι θα είναι κατώτερο προ το ποσό σε σχέση με αυτό που πρότεινε η Κομισιόν, είναι ένα προπολογισμό που εξακολουθεί να διέπεται από μια φιλοσοφία και από μια στρατηγική. Ο προπολογισμό ε, λοιπόν θα καταρτιστεί σε επίπεδο χαμηλότερο από την πρόταση τη Κομισιόν. Βέβαια, γύρω από το τραπέζι νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιοι που θέλουν ε, ακόμη μεγαλύτερη περικοπή. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όμω, τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση για το επίπεδο, νομίζω ότι κανένα δεν θέλει να, να υπερβούμε ε, τις περικοπές που δυστυχώς χρειάστηκε να προτείνω. Υπερασπίστηκα λοιπόν έναν υπερπολογισμό που παρά τα αυτά περιλαμβάνει μια στρατηγική και μια φιλοσοφία και εξακολουθώ να αναζητώ λύση μια λύση η οποία θα προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ της ε, σταθερότητας ε, και της αλληλεγγύης, όπως προείπα, διότι η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται, δράζεται στην αλληλεγγύη. Χωρίς αλληλεγγύη δεν υπάρχει Ένωση. Και νομίζω ότι ό,τι έχει να κάνει με τη συνοχή, ε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτά είναι αλληλεγγύη, αλλά δεν μιλάμε για μια μεταφορά μεταφορά πίστος γίνεται όταν δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Εδώ όμως υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις και αυτό το αντάλλαγμα είναι οι επενδύσεις. Επομένως η αλληλεγγύη πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ το τι θα πει απλά μεταφέρουμε κάποιους πόρους που δεν ισχύει για το συγκεκριμένο προπολογισμό και διάκριση επαναλαμβάνω από αυτό που θα ε, σημάνει την παροχή βοήθειας για κάποιους που σημαίνουν κάποια υστέρηση στην κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη αλλά που επενδύουν για να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο της αλληλεγγύης θα πρέπει να το διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο που να μπορούμε να το υπερασπιστούμε. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής εξυγίανσης αλλά και της ανάπτυξης. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δεν μπορούμε να συνάψουμε ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη τον Ιούνιο και μετά μετά από κάποιε εβδομάδε, μετά από κάποιου μήνε να υιοθετήσουμε έναν προεπλισμό που οδηγεί προ την αντίθετη κατεύθυνση. Άρα πρέπει να προσπίσουμε τη στρατηγική και τη φιλοσοφία αυτή. Έχουμε τη στρατηγική 2020 και το έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια του πρώτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο διοργάνωσα το Φεβρουάριο του 2010. Επομένω. εγώ θα διατηρήσω την ισορροπία, θα την υπερασπιστώ. Φυσικά και θα πρέπει να συμφωνήσουν μαζί μου 27 χωρίς μέλη. Φυσικά και το Κοινοβούλιο. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Και το είπε και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι συζητήσει που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και για να υπάρξει αυτή η ισορροπία, να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, πρέπει να σα πω ότι είμαι ο μόνο που την προσπίζουμε. Φυσικά έχω στο πλευρό μου τον πρόεδρο τη Κομισιόν. Δεν θα λάβει αυτό όμω την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα, την τελική έκβαση. Αντίθετα από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω, παραλαμβάνω είμαι ο μόνο ο οποίο αυτή την ισορροπία και πρέπει να το γνωρίζετε. Συμφωνώ επίση με όσους έκαναν μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και νομίζω ότι είχα κάνει και εγώ αυτή την παρατήρηση όταν ήταν πρωθυπουργό ο κύριος ε, Φερχόφστατ και ενημέρουν το Γλυκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου τότε. Είναι ένας προπολογισμό που συζητάμε που είναι γύρω στο 1% του ΑΕΠ. Και συζητάμε μέχρι σε σχάτων, θα έλεγα, αυτό το 0,1-0,2% του ΑΕΠ δεν ξέρω, για να ενθουσιαστώ ε, μου χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ε, και θα πρέπει κάπως να σχετικοποιήσουμε και να αποδραματοποιήσουμε την κατάσταση. Σίγουρα λύση πρέπει να βρούμε. Και θα κάνω κάθε ε, προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ούτε και να υπαταλπιστεύουμε και να υπερβάλλουμε πρέπει. να μην γελιοποιούμε τα πράγματα. Έχουμε τους καθαρούς εισφορείς από τη μία και τους αποδέκτες πόρων ε, από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Net recipients, net contributors. Και λέτε ότι υπήρξε αντιπαράθεση. Δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Μην φτάσουμε λοιπόν να γελοποιούμε τα πράγματα και να δημιουργούμε μία μονήρη αντιπαράθεση μεταξύ φτωχών πλουσίων. Σε καμία περίπτωση δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Ούτε επίση θα πρέπει να παρουσιάζουμε τη συζήτηση σαν να είχαμε 27 που υποστήριζαν τα εθνικά του συμφέροντα και έναν ή δύο που και δεν ήταν και συνέχεια με στην αίθουσα, που πρόσπιζαν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και πάλι η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη από αυτό. Φυσικά, όταν κάποιο είναι πρόεδρο ή πρωθυπουργό τη χώρα του, φυσικά και πρέπει να προασπίσει τα εθνικά του συμφέροντα, έτσι δεν είναι. Ή να ε, απαγορεύεται να προσπίσει κανεί τα εθνικά συμφέροντα. Όχι. Αλλά σίγουρα πρέπει να ενταχθεί μέσα σε ένα ε, γενικότερο σχέδιο και όραμα. Ο ρόλο λοιπόν του Πρόεδρου, του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να υπενθυμίσει όσου θέλουν να ξεχάσουν ότι έχουν και ευρωπαϊκά συμφέροντα, που δεν το ξεχνάνε όλοι σε καμία περίπτωση, αλλά καθήκον μας είναι να του το υπενθυμίζουμε τέλο πάντων. Δεν υπάρχουν 27 εγωιστές γύρω από το τραπέζι. Και έξω από την αίθουσα είναι όλοι γενναιόδοροι. Πάλι και αυτό η είναι ε, και αρνούμε ε, να διαβώ αυτό το δρόμο. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη πραγματικότητα. Αγαπητοί βουλευτές, κάποιοι ε, ουσιαστικά με στριμώξε στον τοίχο και μου λέτε ότι πρέπει να έρθω στο επίπεδο, στο ύψο των ιδρυτών πατέρων. Εγώ αυτό που πρέπει να κάνω είναι να καταρτήσω προπολισμό για την περίοδο 2014-2020 που θα διέπεται από τον, ε, όλη στρατηγική και φιλοσοφία ε, που δείπε και την πρόταση της Κομισιόν. αλλά ότι ουσιαστικά ε, είμαι ε, ο υπηρέτηση, ακολουθώ τις επιταγές των μεγάλων χωρών που μπορεί να με κατηγορήσετε και είναι εσφαλμένο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όλοι αντίθετα. Ε, τους έχω όλους απέναντί μου, πρέπει να σας πω. Όλοι είναι αντίθετοι με αυτά που λέω. Και παρόλα αυτά θα κάνω ό,τι μπορώ για να βρω μια ισορροπημένη λύση η οποία θα λαμβάνει κατά το δυνατόν υπόψη τις επιθυμίες και τα μέλήματά σας, ίσως δεν θα είναι ένα συμβιβασμός, ε, όπως κανείς μπορεί να τον σχεδιάσει, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα είναι ένας ε, ανεκτός συμβιβασμός που θα μπορεί κανείς να τον αποδεχθεί και θα πρέπει να δώσετε και εσείς τη συγκατάθεσή σας, τη συνένεσή σας, γιατί αλλιώ θα είναι φρούδες οι προσπάθειες που θα έχουμε καταβάλει μέχρι τώρα και μάτες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μάρτιν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, και ο Σαούλ έγινε Παύλος. Οπότε μπορώ να ε, επαναλάβω την ε, έκκλησή μου γιατί έχουμε τέτοια δυσπισία προς τον πολίτη ότι ε, θεωρούμε ότι υπάρχει τέτοιο έλλειμμα διότι και εσείς κύριε Μπαρόζο δυστυχώς το ίδιο σκέπτεστε το θέμα είναι ε, γιατί απορρίπτεται την κριτική και δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, αν δεν μπορέσει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σχετικά ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν σχολιάσατε τη σύγκληση εθνοσυνέλευσης και μόνο εάν μπορέσει κανείς να συνδυάσει την δημοκρατία συστηματική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον αγώνα κατά των χρηματαγορών που θα κερδίσουμε το χρόνο για να καλύψουμε το ε, χαμένο χρόνο μέχρι τώρα. Κύριε Βαν είπαμε ότι ενδέχεται να υπάρξει ένα συμβιβασμό στο τέλος τον οποίο πρέπει να αποδεχθούμε. Σας επαναλαμβάνω και πάλι, ο συμβιβασμός θα είναι κακός και ο κάθε κακός συμβιβασμός θα εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα αίσιο περαιτέρω μέλλον. Δεν θα το στηρίξουμε εάν υπάρχει κατακαιρματισμός. Δεν θα στηρίξουμε τη θέση αυτή και γι' αυτό σας παρακαλώ να καταλήξετε σε μία συμφωνία η οποία επίσης θα μπορέσει εδώ να γίνει αποδεκτή διότι δεν πρέπει η ε, υπεύθυνοι να μιλούν με δύο γλώσσες, μία εδώ και μία στις χώρες τους. Θα πρέπει ε, όλοι να φροντίσουν οι ε, πολίτες να μην εμπλακούν σε μία διαμάχη για την οποία δεν ευθύνονται και όπου υπάρχει απλώς σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Αυτό ε, δεν θα μπορέσουμε να το δεχτούμε και δεν μπορούμε να είμαστε επικοδομητικοί σε μια τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Ανδρέασεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μπαγόζο ότι τον ε, ανησύησε πολύ ότι γίνεται εκτός των ε, ε, συνεδριάσεων. Ό,τι δεν σας αρέσει λέτε ότι είναι λαϊκίστικο. Νομίζω ότι όπως είπε και ο κύριος Βανροπόη, θα πρέπει να αποφύγετε και κάποια σχόλια. Τα γεγονότα δεν είναι λαϊκίστικα σχόλια. Ίσως με κάποιους είσαστε πολύ γενναιόδοροι. Αυτή τη στιγμή δεν, ε, και οι πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας είδαν ότι δεν πηγαίνουν σωστά τα χρήματα και θέλουν περισσότερο πόλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και η Διακομισιό το έκανε. Επιτρέψαμε σε αυτά τα κονδύλια να πάνε εκεί που πήγαν και οι άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα διότι και οι ίδιοι υποφέρουν από τις περικοπές. Οι ίδιοι πόροι δεν είναι κάτι που θα ε, βελτιώσουν το πρόγραμμα, θα το επιδεινώσουν διότι ε, αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι χειρότερη κατάσταση και θα ξεφύγει από τα χέρια μας και όλη η ουσία της διαπραγμάτευσης. Ευχαριστώ κύριο Τσάραντιλ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπαρόζο, ο οποίος είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η καταπολέμηση της διαφθοράς. Νομίζω ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά Είπατε πολλές φορές ε, ότι ε, πολλές φορές οι συζητήσεις αναγάγονται μόνο στο ιδεολογικό στοιχείο. Συμφωνώ μαζί σας. Και πολύ συχνά πρέπει να τονίζουμε ότι αυτό το πράγμα είναι αμφίδρομο. Δηλαδή κάποιος μιλάει κάποια φορά ε, με σαφήνεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος άλλος μοιράει πιο φεντραλιστικά, Κάποιο κάνει τέτοιου είδους ε, ε, σχόλια και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απορρίψουμε γιατί είναι ακραίο. Κύριε Βον Ρομπάι, εκτιμώ πάρα πολύ τον ε, τόνο με τον οποίο κάνατε εσείς και το ύφος στα σχόλια σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εύχομαι και επιθυμώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριφερθεί όρημα και σοφά ώστε να μην μπλοκάρει την όλη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κονμπεντίτ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όταν έχουμε αντίθετες απόψεις δεν σημαίνει ότι είναι θέμα ιδεολογικό, απλά θέλουμε μια άλλη Ευρώπη. Την Ευρώπη που θέλετε εσείς δεν τη θέλουμε εμείς. Είναι πολύ απλό. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μη μας ζαλίζετε. Δεύτερον, Δύο πράγματα κατάλαβα εγώ. Το πρώτο, ότι υπάρχουν πολλές κόκκινες γραμμές. Για μας, για παράδειγμα, προπολογισμό της Κομισιόν. Και έπειτα, στο εσωτερικό της δομής, η δομή δηλαδή, αν δεν έχουμε την ετήσια ιστορική ευελιξία. Αυτοί λένε όχι. Εάν δεν υπάρχει η αναθεώρηση μετά από δυόμιση χρόνια, αυτοί λένε όχι. Άρα, πάρτε το αυτό, είναι οι κόκκινες γραμμές του Κοινοβουλίου. Αυτοί οι άλλοι και εμείς πλειοψηφία. Ούτε τα τρία πέμπτα θα έχετε. Λοιπόν, το ξέρετε ήδη. Πείτε στι κυβερνήσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν δεν έχουμε το τάδε, το δίνα, το τρίτο, θα πει όχι το κοινοβούλιο. Και έτσι θα ε, προχωρήσουμε λιγάκι. Κάποιε φορέ, ξέρετε, τα πράγματα είναι απλά, με τα λέμε και απλά. Ευχαριστώ. Πολλέ φορέ για να επιτύχει μία συμφωνία θα πρέπει να πούμε τι υπάρχει εντός και όχι τι δεν υπάρχει. Δηλαδή στην πολιτική για να η συμφωνία θέλουμε να προσθέσουμε κάποια στιγμή. Τώρα έχουμε τρία στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα η ρήτρα της αναθεώρησης. Σωστά είπε ο κύριος Λαμασού ότι θα πρέπει να έχει μια τέτοια γενική ρήτρα αναθεώρησης που υπήρχε στο αρχικό κείμενο και αντικαταστάθηκε με κάτι που αφορά μόνο το Ταμείο συνοχή. Δεν είναι σωστά έτσι τα πράγματα. Πρώτο στοιχείο ήταν αυτό. Δεύτερον, οι ίδιοι πόροι. Αυτή τη στιγμή οι πραγματικοί ίδιοι πόροι είναι αυτοί που συλλέγονται από τα κράτη-μέλη και μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το πράγμα θα έπρεπε να είναι αντίθετα. Η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει το FTT και να μεταφέρει ένα μέρος αυτού του φόρου στα κράτη-μέρη. Τρίτον, η ευελιξία. Η ευελιξία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόσο σημαντική όσο και τα κονδύλια και τα ποσά. Δεν συμπεριλαμβάνει το κείμενο. Ευελιξία μεταξύ των διαφόρων κεφαλαίων και μεταξύ των διαφόρων ετών. Σε αυτά λοιπόν τα τρία στοιχεία πιστεύω την ευελιξία, όχι τα κείμενα, τις πραγματικούς ίδιους πόρους, δηλαδή δίδοντας έναν ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να του συλλέξει και στην ρήτρα που αναθεώρησες που ανέφερα έχουμε τα κλειδιά για μια δυνατή συμφωνία για αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ για μιση λεπτά ο κύριος Κάουφεν. Κύριε Πρόεδρε, ε, σας εκτιμώ ε, όλοι επιζητούμε τον ίδιο στόχο και θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι για να μπορέσει να πετύχει η δουλειά σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτησή μας, αλλά αυτά τα τελευταία που διαβάσατε δεν αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Ε, συγκρίνεται τον προϋπολογισμό με αυτόν ο οποίος είχε υιοθετηθεί το 2006 το οποίο σημαίνει ότι το 2014 θα υπάρχει μία ε, ισχυρή περικοπή σε αυτά τα πακέτα πράγμα το οποίο θα είναι αντιπαραγωγικό. Είναι χρήματα που πηγαίνουν στις περιφέρειες. Δεύτερον, είπατε ότι υπάρχει μία μικρή αύξηση στην έρευνα και καινοτομία. Τα τελευταία 7 χρόνια η Ευρώπη υποχωρεί. Δηλαδή χάνουμε την ταχύτητα που είχαμε. Και αν υπάρξει μία μικρή αύξηση, οι ε, ανταγωνιστές μας οι οποίοι επενδύουν περισσότερο περισσότερο στην έρευνα και τεχνολογία θα μπορέσει να καλύψει το κενό. Διαφορετικά το κενό αυτό θα αυξάνεται και το 2020 θα είναι ένα μεγάλο χάσμα και δεν μας ικανοποιεί. Ζητάμε έναν ισοσχελισμένο προϋπολογισμό. Βλέπουμε όμως ότι τα κράτη θέλουν να δεχθούν οτιδήποτε αρκεί να υπάρχει περικοπή του προϋπολογισμού. Ούτε αύξηση της διαφανείας ούτε τίποτα. Οπότε δεν καταλαβαίνω το θέμα για τις εκτόσεις. Όλοι κάνουν συμβιβασμίους είπατε, αλλά μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Αλλά οι συμβιβασμοί ε, κινείται προς τα λίγα κράτη που είναι αμετακίνητα και πάλι μιλάμε για εκτόσεις. Μιλάμε ε, για δώρα σε κράτη-μέλη που δεν επιτρέπουν στο σύστημα να λειτουργήσει. Υπάρχει η έλλειψη ευελιξίας ακόμη και στην μεσοπρόθεσμη προσαρμογή και τέλος ε, το ενιαίος χαρακτήρας του προπολογισμού γιατί εάν όλες οι προσπάθειες είναι για να μειωθεί ο προϋπολογισμός και όχι για να υπάρχει ένας άλλος προπολογισμό, πώς θα τον χρηματοδοτήσουμε. Εξού και ζητάμε να έχουμε μία ευρεία εικόνα διότι αυτές είναι οι προτεραιότητες και ε, θα μπορέσει έτσι να είναι πιο αποτελεσματικός ο προϋπολογισμός και να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες. Όταν είχαμε συναντηθεί με τον επικεφαλή του επιτελείου σας μας είχε πει ότι αυτή είναι η προσγείωση αλλά υπάρχει μία περιοχή no-fly zone όπου απαγορεύονται οι πτήσεις πάνω από το κοινοβούλιο και πρέπει να συνδυαστούν τα δύο. Και τώρα ο κύριος Μπέγκη για 4,5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κάλφιν, ο οποίος είναι συνεισηγητής και εγώ ε, συμφωνούμε πλήρως. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχουν γρήγορες διαπραγματεύσεις που να καταλέξουν σε ένα αποτέλεσμα, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Οι συζητήσεις με ε, την Προεδρία είναι πιλωτικά προγράμματα, τα briefing, debriefing και μέχρι στιγμής ήταν επικοδομητικά. Αλλά τώρα δεν βλέπουμε να υπάρχει συνέχεια. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα θεσμικά όργανα όπως προβλέπουν οι συνθήκες ε, ε, πρέπει να ε, λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να υιοθετηθεί το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Και πρέπει να σας πω ότι ανησυχούμε πώς θα γίνει αυτό. Ε, ε, δεν θέλουμε να υπάρχει κρίση αλλά η μη συμφωνία δεν σημαίνει καμία κρίση σημαίνει χειρισμός των αριθμών μια κακή συμφωνία η οποία δεν ε, υιοθετεί επαρκώς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι καλή και θα πρέπει να μας ακολουθήσει και το Συμβούλιο και να γνωρίζει σαφώς περί τίνος πρόκειται και σας είπα ποια είναι τα ψηλές δαπάνες. Ε, οι δαπάνες ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη εις ε, τους, εις τους εθνικούς προϋπολογισμούς που είναι εθνισυγενείς και πρέπει να υπάρξουν προσφορές, να τις συζητήσουμε μαζί, να μην μπλοκάρουμε την πρόοδο και κάποια στιγμή το Συμβούλιο θα χρειαστεί να αναγνωρίσει αν συνεχίζει έτσι να χρησιμοποιεί τους αριθμούς ποιες ε, είναι οι δραστηριότητες οι οποίες θα καταργηθούν αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση και που έχουν, έχουμε αποφασίσει. Για να δούμε πώς κόστησαν εν τη σοφία τους αυτά τα οποία αποφάσισαν στο Συμβούλιο εδώ και 10 χρόνια ε, και πού οδήγησαν κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Σας συζητάμε για ένα πακέτο. Όσο πιο δύσκολοι είναι οι αριθμοί, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε γενική ευελιξία και όχι contingency margin χρειαζόμαστε μία δέσμευση ότι θα γίνει σεφαστός ο προϋπολογισμός και όχι ε, η διασπάθηση του προϋπολογισμού. Θα χρειαστούν συγκεκριμένα μέτρα και όχι την review που είχατε δεχθεί την προηγούμενη φορά και θα πρέπει ε, να μπορέσει κανείς ε, να προχωρήσει εις ε, την στην εφαρμογή του προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πάντοτε και πρέπει να εφαρμοστούν και τα πολυετή προγράμματα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, θα εμπλέξετε το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αν διαβάσω το blog σας, βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα προχωρήσει σε νομοθετική πορεία αλλά μετά διαβάζω ότι ο προϋπολογισμός για την περίοδο μέχρι το 2020 θα υιοθετηθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλύτερα θα ήταν να γράφει κανείς τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι μετά από συνένωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πλειοψηφική υπερψήφιση θα μπορέσει ομόφωνα να αποφασίσει το Συμβούλιο. Άρα θα πρέπει αυτή τη στιγμή να σεβαστείτε τις ευαισθησίες μας, να κάνετε τις διαπραγματεύσεις κατά τρόπον ώστε στο τέλος να μας φέρετε μία πρόταση για τη διαθεσμική συμφωνία την οποία θα μπορέσουμε και εμείς να προωθήσουμε στην Ολομέλεια με θετικό πρόσημο διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη εάν δεν υπάρχει μία σωστή συναλλαγή μαζί μας. Και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Παρακαλώ να σεβαστείτε αυτό το οποίο προβλέπει η συνθήκη για τον πρόεδρο των θεσμικών οργάνων και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε απλές λύσεις για να προχωρήσουν. Θα σας στηρίξουμε αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα και δεν είναι εύκολο να προσπαθήσει κανείς να επιτύχει υπερψήφιση στην Ολομέλεια, άρα πρέπει πρέπει και εσείς να μας βοηθήσετε και σας ευχαριστώ. Ωραία. Νομίζω ότι τώρα είναι, ε, είναι σκόπιμο όπως ζητά η συνθήκη να κηρύξω τη λύση της ε, συνεδριάσεως ευχαριστώντας τον πρόεδρο Βαν και τον κύριο Μπαρόζο.